Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Πριν από αυτό έχει ζητήσει το λόγο για point of order ο κύριος Αχματ Μπασίρ. Παρακαλώ κύριε Μπασίρ, έχετε το λόγο. Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ να ακούσουμε τον κύριο Αχματ Μπασίρ.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 It's a, it's honorable chair. Αξιότιμε πρόεδρε. Χθες στο Sky News είδαμε είδε όλος ο κόσμος